ladies and gentlemen, I think we should... Κυρίες και κύριοι, νομίζω πως θα πρέπει να ξεκινήσουμε. Further, I will speak... Και θα συνεχίσω στα γερμανικά, οπότε θα ήθελα να σας ζητήσω να βάλετε τα ακουστικά σας, εάν δεν γνωρίζετε τη γερμανική. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητοί προσκεκλημένοι μας, Χαίρομαι ιδιαίτερα ε, για το γεγονό ότι μπορώ να σας ε, καλωσορίσω σήμερα και σε αυτό το πάνελ εκ μέρους ε, και της Επιτροπής Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο τουρισμός και ο πολιτισμός, ειδικότερα στην Ευρώπη, συνδέονται στενά μεταξύ τους, ειδικότερα λόγω της πλούσιας πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Και γι' αυτόν τον λόγο και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκαταλέγονται στους, στο στους κύριους προορισμούς παγκοσμίως του τουρισμού. Και η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί ακριβώς αυτό τον συνδετικό ε, κρίκο μεταξύ των κατώμελων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μεταξύ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων περιοχών της, ε, ε, του κόσμου. Και ακριβώς για να ανταποκριθούμε, για να αποκριθούμε σε αυτόν τον σε αυτή τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέλεξαν το επόμενο έτος ως το Ευρωπαϊκό έτος της πολιτιστικής κληρονομιάς και ο στόχος είναι να καταστεί πιο γνωστή αυτή η πολιτιστική κληρονομιά, να υπάρχει μεγαλύτερη διαπολιτισμική κατανόηση ε, και να υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για μια Ευρώπη η οποία θα είναι απτή για τον τουρίστα. Και αυτό βέβαια θα μπορούσε πάντοτε να συνοδεύεται ακριβώς από τα ταξίδια και από τον τουρισμό ταυτόχρονα. Και το 2018 δεν θα είναι μόνο το ευρωπαϊκό έτος της ε, πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και το έτος τουρισμού Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και Κίνας. Η προώθηση του τουρισμού ανάμεσα σε αυτές τις δύο ε, περιφέρειες του κόσμου θα επιτρέψει στους πολίτες τους να γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους. Και εδώ, σε αυτό το επίπεδο, η πολιτιστική κληρονομιά θα παίξει αποφασιστικό ρόλο. Ο πολιτισμός είναι και θα παραμείνει και στο μέλλον ένας από τους κύριους μαγνήτες εντός εισαγωγικών του τουρισμού. Αλλά ε, σε ορισμένε περιπτώσει ε, δεν υπάρχει πάντα συνέργεια με τον τουρισμό. Για παράδειγμα, ε, βλέπουμε πω ήδη σε ορισμένε περιοχέ ο τουρισμό να έχει και αρνητικό αντίκτυπο. Για παράδειγμα, οι τεράστια αριθμοί τουριστών που καταφτάνουν σε κάποια νότια σημεία δημιουργεί πλέον και ανησυχίε. Για παράδειγμα, ε, οι 56.000 ε, κάτοικοι της ε, παλιάς πόλης της Βενετίας βρίσκονται αντιμέτωποι με 30 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως. Ε, και η ζωή στις παλαιές πόλεις, ε, στις παλιές γειτονίες ορισμένων ευρωπαϊκών ε, πόλεων δυσκολεύεται από τους τουρίστες, από διάφορους δηλαδή νέους οι οποίοι φωνάζουν και διάφορους οι οποίοι κουβαλάν selfie sticks. Κάποιοι δηλαδή κάτοικοι αυτών των παλαιών πόλεων δεν μπορούν πλέον να ανταποκριθούν ούτε στις τιμές των νοικιών, ούτε και στις τιμές των εστιατορίων και των μπαλ. Και ε, ταυτόχρονα γίνεται συχνά και λόγος για ένα είδος τουριστικοποίησης, ε, το οποίο δηλαδή σχετίζεται ε, και με τις δράσεις του εξοραϊσμού. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά με αυτήν την τουριστικοποίηση ότι διαταράσσεται τόσο πολύ ο κοινωνικός ιστός που να έχει μετατραπεί τελείωσε. Ε, και χαίρομαι ιδιαίτερα το γεγονό που μα προσκάλεσε ε, ο πρόεδρο Σταγιάννη να κάνουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα. Γιατί πραγματικά έχει νόημα ε, να γίνει αυτή η συζήτηση προκειμένου να προωθηθεί η Ευρώπη ω τουριστικό προορισμό. Γιατί αυτό μα επιτρέπει να έχουμε ένα καλύτερο διαπολιτισμικό διάλογο με τη Γίνα και καλύτερη προώθηση των σύστημα. αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί και ε, θετικά ε, ερεθίσματα για την οικονομία. Όμω, για την προώθηση του τουρισμού στην Ευρώπη θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μα επιγόντω και δύο ακόμα διαστάσει. Τη βιωσιμότητα και την ανάληψη τη ευθύνη, την υπευθυνότητα. Και θα ήθελα ε, μετά από αυτά τα λόγια να δώσω το λόγο στους 15 προσκεκλημένους μιλητές μας, τους οποίους καλωσορίζω θερμά. Όλοι σας θα έχετε κατά το μέγιστο τέσσερα λεπτά στη διάθεσή σας ε, χρόνο αγόρευσης και αν γίνεται τρία λεπτά και πραγματικά σας ε, καλώ επίμονα να τηρήσετε αυτό το χρόνο αγόρευσης και να μην θυμώσετε εάν σας διακόψω σε περίπτωση που ξεπεράσετε αυτό το χρόνο αγόρευσης. Ε, πρόκειται δηλαδή και για δικαιοσύνη, να προσπαθήσουμε δηλαδή να διασφαλίσουμε τον απαραίτητο χρόνο αγόρευσης για όλους τους ομιλητές που θα ακολουθήσουν τον καθένα από εσά και ίσως στο τέλος να μας μείνει και λίγος ο χρόνος για να συζητήσουμε. Να σας ενημερώσω επίσης ότι θα υπάρξει web streaming αυτή της ε, συνεδρίασης, δηλαδή μετάδοση online και μπορείτε να την παρακολουθήσετε και από τον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μπορείτε να παρακολουθήσετε ε, την συνεδρίαση σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ευχαριστώ και τους διερμηνείς οι οποίοι θα διευκολύνουν το έργο μας και στη σημερινή μας ε, διάσκεψη. Αν θέλετε να διαβιβάσετε κάποιο μήνυμα μέσω ε, Twitter μπορείτε να το κάνετε μέσω του hashtag tourismus.eu. Ε, αναμένω λοιπόν με μεγάλο ενδιαφέρον τη συζήτηση που ακολουθήσει και ε, πρώτος ομιλητής είναι ο Δήμαρχος της Βενετίας, ο κύριος Μπρουνιάρο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο Ταγιάννη που με κάλεσε να εκπροσωπήσω την πόλη της Βενετίας σε αυτή τη σημαντική εκδήλωση. Χαιρετίζω την κυρία Ειρήνα Μπουκόβα που είναι πρόεδρος και διευθύντρια, μάλλον η διευθύντρια, γενική διευθύντρια της UNESCO που όπως είπε θέλει να δώσει απαντήσεις σε περίπλοκες, σε περίπλοκα προβλήματα. Λέγαμε λοιπόν ποια είναι η αξία του τουρισμού. Θέλω να το υπογραμμίσω. Είναι μια αξία τουρισμός διότι ε, έχουμε πρόσωπα, άτομα, είμαστε άτομα Υπάρχουν άτομα που έρχονται στη Βενετία Φερρυπίν, που αγαπούν την πόλη και γι' αυτό ξεκινήσαμε μια εκστρατεία για σεβασμό, λέγεται σεβασμός για τη Βενετία, διότι ζητούμε κάτι μην την, να μην καταστραφεί και να τη σέβονται. Το πρώτο μέτρο που επεξεργαστήκαμε, κατασκευάσαμε μαζί με την Ιταλική κυβέρνηση και την UNESCO, την UNESCO την ίδια, βάλαμε μέτρα, μέτρα ενημέρωσης. Θέλουμε να ενημερώσουμε τους διάφορους ε, διάφορες εταιρείε και αυτούς που έρχονται στις διάφορες γλώσσες για να μπορούν για να σέβεστε, να σέβονται τους κανόνες που τους καταλαβαίνουν. Υπάρχουν βέβαια και εμπόδια και δυσκολίες κάποιες ε, ημέρες και κάποιες εχμές αν θέλετε όταν υπάρχει κακοκαιρία στις ε, παραλίες και λοιπά το καλοκαίρι ε, και έχουμε απρόβλεπτες ακμές, περισσότερο κόσμο και γι' αυτό έχουμε ένα κέντρο στην πόλη, κέντρο ελέγχου, κέντρο ελέγχου όπως δημιουργήθηκε και στη Νέα Υόρκη που αφορά την ασφάλεια, την αστυνόμευση, ε, το, γενικά τη διαβίωση στην πόλη. Λοιπόν, ποιο είναι το μήνυμα που μπορώ να σας δώσω σε τέσσερα μήνα και θα είμαι ακριβώς ε, σε αυτό το περιθώριο το χρονικό που τίθεται. Πρέπει να πω λοιπόν ότι πρέπει να εξηγήσουμε τη δυσκολία να διχειριστούμε μια πόλη. Το να διχειριστεί κανείς μια πόλη όπως είναι η Βενετία, συνεπάγεται κόστος απίστευτα υψηλό όσον αφορά ε, βιωσιμότητα κλπ, αστυνόμευση κλπ και καθαριότητα. Αγαπούμε τους ανθρώπους, είμαστε ικανοποιημένοι που έρχονται επισκέπτε στη Βενετία και γι' αυτό το μήνυμα που θα πρέπει να καταφτάσει. Λαμβάνοντας υπόψη τη 19 Ιανουαρίου που θα γίνει μεγάλη εκδήλωση και θα συμμετάσχουν οι διάφορες τουριστικές εταιρείες της Ευρωπαϊκής Ενώσεω και τη Κίνα, διότι έχει ενταχθεί πλήρω η Βενετία στι μεγάλε διαδρομέ ε, τη διαδρομή του μεταξιού. Χαιρόμαστε να φιλοξενούμε του φίλου του Κινέζου. Έχουμε άριστη συνεργασία και όσον αφορά τον πολιτισμό και την ιστορία με του Κινέζου. Αλλά πρέπει να αναπτύξουμε ε, και μια περιοχή τη Πόρτα Μπαριέρα, ένα από τα πιο μεγάλα ε, ε περιοχέ που έχει ε, περάσει από κάποια ύφεση και έχουν χαθεί 30.000 θέσει εργασία σε αυτή την περιοχή. Θέλουμε να ξαναπροωθήσουμε και την κατασκευή, τη βιομηχανία και την λιμενική, την, την περιοχή του λιμένου και ε, διάφορα άλλα συναφή επαγγελμάτα και να μειώσουμε τις τουριστικές πιέσεις κατά κάποιο τρόπο που μπορεί να έχουν αρνητική συνέπεια για την πόλη. Λοιπόν, εκεί που ήταν κάποια εργοστάσια υπήρχαν στην πρώτη μπαριέρα, ε, θέλουμε αυτό να αντιμετωπίσουμε για να λάβουμε υπόψη και τις πιέσεις που ασκήσει το τουριστικό ρεύμα. Μπορεί να χρήσιμη αυτή η εμπειρία μας και σε διάφορες άλλες πόλεις. Αυτό που ξεκινούμε να κάνουμε θα το συζητήσουμε με τη διεθνή κοινότητα και το συζητούμε πάντα. Και τελευταία είδηση που δίδω, ε, πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι, η κυβέρνηση θα κάνει τη δήλωση, ευχαριστώ γι' αυτό, ότι τα, τα πλοία, η κυκλοφορία αυτή η περίφημα, ε, δεν θα περνάνε τα κρουζεροπλία μπροστά από τον Άγιο Μάρκο, θα κάνουν άλλο γύρο. Ε, δεν θα περνάνε μέσω από ε, το καναλιού που είναι μπροστά από την Τζουντέκα. Ε, λοιπόν, ευχαριστούμε για τις προσκλήσεις ε, και που μας καλούν από τη διεθνή κοινότητα. Είμαστε κοντά, εμείς θα προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε μέτρα βιωσιμότητας και μετά θα περιγράψουμε και στους άλλους αυτά τα μέτρα που ίσως και κάποιοι άλλοι να χρειάζονται παρόμοια μέτρα όπως εμείς. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ και για την απόλυτη τήρηση του χρόνου σας. Επόμενη ομιλήτρια είναι η Αντιδήμαρχος της Βουδαπέστης, η κυρία Σάλαϊ Ντομπροβίνσκι και ελπίζω να μην το κατακρεωργώ. Thank you very much. So... Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε. Ως Αντιδήμαρχος της Βουδαπέστης θα ήθελα να σας πω δύο λόγια ε, για το τουριστικό προορισμό Ευρώπη. Όλο και περισσότερο πόλεις ε, συμμετέχουν ε, στη δημιουργία ενός σήματος, μιας, σήματος κατατεθέντος, branding και προσπαθούν να δώσουν σε ένα διεθνές στερέωμα μια ταυτότητα στην πόλη τους και στον τόπο τους. Αυτό τι σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε τοπικές ταυτότητες, ε, προβολή μιας πόλης, αλλά αυτό δεν μπορεί να κατασκευαστεί σε ένα εργαστήριο ως αμάρκα. Δεν μπορεί να είναι τεχνητό και κατασκευασμένο θα πρέπει να υπάρχει ταυτότητα που να τροφοδοτείται από τους πολίτες, από ε, ε, εμβληματικές πρωτοβουλίες και από τη ζωή της πόλης. Και δεν είναι μόνο μια εικόνα αυτό το branding, είναι και ένα μονοπάτι προς το μέλλον. Ε, και θα πρέπει σε αυτό το κοκτέιλ να μπει και η ζωή των πολιτών και η επιθυμία των καθημερινών πολιτών, ακόμα καλύτερα. Ε, τούτες τις μέρες ε, γίνεται μια προσπάθεια. Ε, εγώ δεν θέλω να σας κουράσω με κοινοτοπίες και να σας κάνω να βαρεθείτε. Απλώς ο κόσμος αλλάζει και θα πρέπει να το καταλάβουμε, να το κατανοήσουμε και να καθορίσουμε την κατεύθυνση των αλλαγών αυτών. Ε, οπότε δεν είναι ντροπή να μάθουμε από κάποιους που έχουν με επιτυχία περάσει αυτές τις σχολίες και τις έχουν ξεπεράσει. Όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος προηγουμένως, θέλω να πω και εγώ ότι όταν μιλούμε για ανάπτυξη ή για το μέλλον, τίθεται ένα ερώτημα που αφορά εκείνους οι οποίοι ζουν στις πόλεις και με ποιο τρόπο ο τουρισμός μπορεί να κάνει τη ζωή στην πόλη πιο βιώσιμη, πιο ε, αηφόρο και πιο ανθρώπινη. Κατάλαβαμε λοιπόν ποια είναι τα καθήκοντα και αποστολή μας. τρόπος είναι με ποιο... Ε, η ερώτηση μάλλον είναι με ποιο τρόπο θα το υλοποιήσουμε αυτό. Ποια είναι η θέση μας, ποιος είναι ο ρόλος μας. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να φύγουμε από τη βολή μας και να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε για το μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Σάλαε. Και τώρα θα ακούσουμε ε, το δήμαρχο της Κωνσταντσα που είναι ένα λιμάνι στη Ρουμανία. Καλωσορίζω θερμά τον κύριο Φαγκαντάου και τον παρακαλώ να μας παρουσιάσει ε, τη ε, δική του τοποθέτηση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Θέλω να σας συγχαρώ καταρχάς τον κύριο Ταγιάννη για αυτή τη σημαντική διοργάνωση και θα ήθελα επίσης να ε, δράξω την ευκαιρία για να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία ε, Τσαπαρντέλ, ε, την Ευρωβουλευτή που μαζί σας κυρία Πρόεδρε ανέλαβε μια πρωτοβουλία για τον τουρισμό και την Ευρώπη. Λοιπόν, είμαι δήμαρχος της Κωνσταντσα, μια πόλη πολύ παλιά, ένα παλιό λιμάνι, τουριστικό, παραμεθόριο και είναι και τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάνω από 300.000 κατοίκους έχουμε και είμαστε γνωστοί λόγω του λιμανιού. Είναι πολύ μεγάλο λιμάνι στον Εύξηνο Πόντο. Και συνδέει την Ευρώπη με τον κόσμο. Αλλά η Κωνσταντσα δεν είναι γνωστή μόνο ως λιμάνι, αλλά και ως τουριστικός προορισμός. Αν σας πω Μαρμάγια μπορεί να σας λέει τίποτα περισσότερο πριν από τέσσερα χρόνια κέρδισε το βραβείο για την πιο δυναμική παραλία, ή μάλλον παραλίες στην Ευρώπη. Μέχρι πρόσφατα ήταν ένα θέρετρο, μικρό, χωριουδάκι, ε, ένας ωραίος προορισμός για καλοκαιρινές διακοπές. Με την υποστήριξη και των ευρωπαϊκών κονδυλίων όταν μπήκαμε στην ευρωπαϊκή οικογένεια καταφέραμε να αναπτύξουμε αυτό το μικρό ε, τουριστικό θέατρο που ήταν απομονωμένο και να το απογειώσουμε. Έχει λάβει μια καινούργια διάσταση και δεν αφορά αυτό μόνο το θερινό τουρισμό. Προσπαθούμε να δώσουμε και μια πολιτιστική διάσταση στον τουρισμό, το είπε και η προλαλήσασα αλλά και η πρόεδρος. Είναι σημαντικό να το καταλαβαίνουν και οι τουρίστες αυτό. Η μαζί με μια Ιταλική πόλη θα γιορτάσει ε, την επέτειο ενός γεγονότος που έγινε πριν από 2.000 χρόνια. Πριν από 2.000 χρόνια ένας συγγραφέας έγραφε πόσο δυστυχισμένος ε, ήταν ε, στην εξορία, στη Μαύρη Θάλασσα και ξεκίνησε μια δράση. Ήταν ένας Ρωμαίος ε, συγγραφέας και σε συνεργασία με τους Ιταλούς ε, δόθηκε μια συναυλία από έναν από τους πιο σημαντικούς βιολιστές του κόσμου. Έπαιξε Βιβάλντι, είχαμε και ε, κλασικό μπαλέτο με Ιάπωνες χορευτές. Και ήρθαν πάνω από 2.000 ε, νέοι ε, γιατί είχε ένα πρωτάθλημα σκακιού. Και μετά είχαμε ένα πρωτάθλημα τριάθλου που ήρθαν κι άλλοι νέοι από παντού, από όλη την Ευρώπη. Άρα λοιπόν ο τουρισμός δεν είναι μόνο ο τουρισμός, είναι και ε, αθλητικές και πολιτιστικές οργανώσεις και με τα ευρωπαϊκά κονδύλια και την υποστήριξή τους καταφέραμε να επιτύχουμε πάρα πολλά και αυτές ε, οι απομονωμένες ε, παραλίες που είναι τουριστικά θέρετρα μπορούν να αναπτυχθούν και να υπάρχει και μια πολιτιστική διάσταση στον τουρισμό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μας και είναι σημαντικό να γίνουμε κι εμείς ένα τμήμα ε, του μεγάλου δικτύου του τουριστικού. Η πόλη μας είναι πάρα πολύ ωραία. Ελάτε όλοι στην Κωνσταντσα να την ανακαλύψετε. Και το Δήμαρχο της Βενετίας προσκαλώ. Έχουμε ε, πραγματικά ε, υποχρέωση να προστατεύσουμε το περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο η πόλη μας ωραία και ολόκληρη η περιοχή και κάτι μοναδικό πολύ κοντά μας είναι το δέλτα του Δούναβη, μια μοναδική ε, περιοχή φυσικού κάλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στρογγυλή τράπεζα αυτή, τη διοργάνωση και από κοινού μπορούμε να προχωρήσουμε και να πείσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είναι περισσότερο από ένας οικονομικός ε, τουρισμός, ε, κάτι που αποδίδει οικονομικά ωφέλη. Και χαίρομαστε πάρα πολύ για την πρωτοβουλία που ε, αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2018 και το κηρύσσει το έτος της Κίνας. Θέλω να ευχαριστήσω και να ξαναπώ και στον Επίτροπο ότι η Ρουμανία και η πόλη μου η Κωνσταντσα θα το γιορτάσουν όπως αρμόζει αυτό το έτος πολιτιστικής κληρονομιάς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Φαγκαντάου. Ο ο μιλητή μα μάλλον χρειάστηκε να ταξιδέψει περισσότερο από όλου ε, του άλλου για να φτάσει σήμερα εδώ. Οπότε καλωσορίζω ιδιαίτερα θερμά τον ε, κύριο Ντάι, ο οποίο είναι ο επικεφαλή ε, τη Κινέζικη Τουριστική Ακαδημία. αναμένω λοιπόν με ενδιαφέρον την παρέμβασή του, αλλά θα πρέπει να σας αναφέρω ότι θα μιλήσει στα κινέζικα ο κύριο Ντάι. Ωστόσο, οι διερμηνεί ε, θα διαβάσουν την ήδη μεταφρασμένη στα αγγλικά ομιλία του από το κείμενο που έχουμε μπροστά του. Οπότε, δίνουμε το λόγο στον κύριο Ντάι. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, σα ε, χαιρετίζω. Ε, το 2004 ε, όταν επισκέφθηκα την Ευρώπη για πρώτη φορά, επισκέφθηκα πρώτα τι ε, Βρυξέλλε και κοίταζα περίεργα τι διάφορε πόλει, αλλά συνάντησα και διάφορου ανθρώπου που με κοίταζαν και εκείνο η περιέργεια. Και ένα πήρε ε, μια στάση ε, καράτε και μου είπε κουνφού. Κουνφού νόμιζε δηλαδή ότι όλοι οι Κινέζοι ξέρουμε ε, πολεμικέ τέχνε. ή νόμιζαν για παράδειγμα ότι είχα μια πλεξούδα πίσω στο κεφάλι μου όπω οι αρχαίοι Κινέζοι. Πάντως από την άλλη πλευρά ε, πολλοί ακαδημαϊκοί και επίσημοι με υποδέχτηκαν ε, θερμά. Για παράδειγμα ο ε, πρόεδρος του Κοινοβουλίου της περιοχής των Βρυξελών με υποδέχτηκε για ένα γεύμα έξι ωρών και ήμουν πραγματικά βαθιά εντυπωσιασμένο από από την πολύ θερμή υποδοχή. Ε, κατά τα τελευταία 13 έτη, υπό τις εκείνες προσπάθειες των κυβερνήσεών μα ε, και των επιχειρήσεών μα, οι ανταλλαγές τουριστικέ μεταξύ ε, των δύο περιοχών είναι γνωστέ για πολύ μεγάλα του επιτεύγματα. Για παράδειγμα, είχαμε τι περισσότερε ανταλλαγέ τουριστικέ μεταξύ Κίνα και Ευρωπαϊκή Ένωση τον τελευταίο καιρό. Μετά από την υπογραφή τη συμφωνία για το καθεστώ συγκεκριμένου προορισμού, ο αριθμός για παράδειγμα, των τουριστών τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην Κίνα το 2006 έφτασε στα 3,1 εκατομμύρια, ενώ αυτό των Κινέζων τουριστών στι ε, ευρωπαϊκέ χώρε έφτασε στα 3,4 εκατομμύρια. Και βέβαια αν συμπεριλάβουμε και του τουρίστε από το Χονγκ Κόνγκ, το Μακάο και την Ταϊβάν, αυτό ο αριθμό ε, των Κινέζων δηλαδή τουριστών θα ήταν ακόμα υψηλότερο. Ε. Ε, και με βάση του πρώτου υπολογισμού, το εισόδημα τη Κίνα από τον τουρισμό φτάνει στα 14,17 δι δολάρια, ενώ αυτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση στα 11,49 δισεκατομμύρια δολάρια. Άρα λοιπόν και οι δύο πλευρέ έχουν υποφεληθεί τα μάλα από την τουριστική ανάπτυξη, τόσο σε ό,τι αφορά την οικονομική ανάπτυξη, όσο σε ό,τι αφορά και την δημιουργία κατά τόπου θέσεων εργασία. Οι ε, Κινέζοι τουρίστε ταξιδεύουν ε, περισσότερο από κάθε άλλη φορά στην Ευρώπη ε, και πέρα από τις, ε, τους παραδοσιακούς προορισμούς όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ισπανία που αποτελούν δηλαδή τους του του επιλογές επισκέπτονται ολόνα και περισσότερο και άλλε ε, χώρε, όπω το Βέλγιο, η Ελβετία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα, η Τουρκία, η Δανία, η Φινλανδία, η Σουηδία, η Αυστρία και η Τσεχική Δημοκρατία. Ε, και επίσης ε, τους βλέπουμε όχι μόνο πλέον στα μεγάλα μετροπολιτικά κέντρα όπως το Παρίσι, η Ρώμη, το Λονδίνο, η Φραγκφούρτη και οι Βρυξέλλες αλλά και σε πολλές ε, μικρότερες ή και μεσαίες πόλεις και επαρχιακές κομοπόλεις. Και τους βλέπουμε βέβαια όχι μόνο στα τοπικά σημεία προορισμού αλλά και σε διάφορους άλλους προορισμούς, για παράδειγμα σε δημόσιους χώρους και να απολαμβάνουν και άλλου χώρου αναψυχή ή να μετακινούνται, για παράδειγμα, με το μετρό ή με άλλα ε, δημόσια ε, μέσα μεταφορά. Και όλοι ε, προσπαθούν να βιώσουν αυτό που λέει και το αρχαίο κινέζικο ρητό, δηλαδή το να διαβάσει κανεί 10.000 ε, βιβλία και να ταξιδέψει 10.000 μίλια. Σήμερα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα έχουν πραγματικά και το καλύτερο σύστημα ε, σύνδεση ε, μεταξύ του σε ό,τι αφορά τι μεταφορέ. Έχουμε 150 αεροπορικέ εταιρείε οι οποίε συνδέουν την Κίνα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και 2.500 πτήσει καθημερινά. Και χάρη στην πρωτοβουλία μία ζώνη, ένας, δρόμος, ε, ε, ε, ένας δρόμος και τη θέση σε λειτουργία των συνδροδρομων κινα Κίνα-Ευρώπη, οι Κινέζοι τουρίστε θα μπορούν να επισκέπτονται στο εγγύ μέλλον την Ευρωπαϊκή Ένωση και με το τρένο. Και υπάρχει και πρακτική συνεργασία στι τηλεπικοινωνίε, καθώ τα τέλη των διεθνών κλήσεων μειώνονται συνεχώ. Και αυτό επιτρέπει στου Κινέζου τουρίστε να έρχονται σε επαφή ευκολότερα με του αγαπημένου και του φίλου του. Η συνεργασία των δύο κλάδων ε, έχει φτάσει πλέον σε ένα νέο ζενήθ ε, χάρη στην ε, επένδυση των κινέζικων επιχειρήσεων όπως η Χάιζιν Γιάνγκ, η Hainan Airline, New Century και Fusion International. Και βέβαια οι Κινέζοι τουρίστε έχουν τον υψηλότερο βαθμό ικανοποίηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν εντυπωσιαστεί από τι υπηρεσίε, τι τουριστικέ υπηρεσίε υψηλή ποιότητα, όπω αυτό αντικατοπτρίζεται και στην έκθεση συνεχού παρακολούθηση από την Κινέζικη Τουριστική Ακαδημία σε ό,τι αφορά το βαθμό ακριβώ ικανοποίησή για παράδειγμα, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2017, σχετική βαθμολογία της ε, τουριστικής ικανοποίηση. στη Γαλλία ήταν στο 79,35, στην Ισπανία στο 78,85, στη Γερμανία στο 78,54, στην Ιταλία στο 77,61 και στο Ηνωμένο Βασίλειο στο 77,38. Ε, όλα αυτά τα νούμερα είναι σαφώ υψηλότερα από το μέσο όρο. Και οι ε, Κινέζοι τουρίστε είναι ιδιαίτερα εικονοποιημένοι από πτυχέ όπω ε, το αστικό περιβάλλον και η μορφολογία, η ε, φυσική οικολογία αλλά και εξωτική κουλτούρα. Ε, σε συνέχεια από εκεί και μετά τις προηγούμενες συνεργασία που είχαμε με την Ελβετία και τη Δανία το επόμενο έτος θα είναι το έτος τουρισμού μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας και νομίζω πως με τις κοινέ προσπάθειες που θα κάνουν οι κυβερνήσεις μας, οι επιχειρήσεις, οι έρευνητές, ε, ε, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και ε, οι εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης, οι ανταλλαγέ τουριστών μεταξύ Κίνα και Ευρωπαϊκή Ένωση θα φτάσουν νέα ύψη. Και θα ήθελα βέβαια να υπάρξει και περισσότερη καλή θέληση από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στου Κινέζου τουρίστε. Θα μπορούσαν δηλαδή τόσο οι κυβερνήσει και τα μέσα ενημέρωση να περάσουν περισσότερο το μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διατεθειμένη να αποδεχθεί την Κίνα που είναι γνωστή για ένα πολιτισμό 5.000 ετών και που προσπαθεί να οικοδομήσει μια σχετικά ευημερούσα κοινωνία. Και στις ε, δημοσιεύσεις που βλέπουμε τη ετήσια έκθεση σε ό,τι αφορά την τουριστική ανάπτυξη ε, ε, σε σχέση με του κινέζου τουρίστε, βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ θετική συσχέτιση, ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ των διμερών διακυβερνητικών σχέσεων και τη επιλογή των τουριστικών προορισμών. Εάν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να ανταποκριθεί σε αυτή την πρωτοβουλία μια ζώνη, ένας δρόμος τη Κίνα και να έχει θετικές διάδραση με την Κίνα στου τομεί όπω το εμπόριο, επενδύσει, η διπλωματία και οι διαπολιτισμικέ ανταλλαγέ, ε, καθώ και με ένα πιο ευνοϊκό ε, καθεστώ ε, θεωρήσεων, σίγουρα οι Κινέζοι τουρίστε θα επιλέγουν ακόμα περισσότερο τις ευρωπαϊκές χώρες ως τους τουριστικούς τους προορισμούς. Επίσης θα ήθελα να υπάρχουν περισσότερες κοινακίδες, περισσότερα συστήματα διερμηνίας, περισσότερες εφημερίδες και άλλα τηλεοπτικά show τα οποία θα είναι διαθέσιμα στην κινέζικη γλώσσα. Η Πρόεδρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ντάι, για την ομιλία σας αυτή και ευχαριστούμε που μας ήρθατε κιόλας και συμμετέχετε σε αυτή τη διάσκεψη. Πριν περάσω στον επόμενο ομιλητή, θα ήθελα να καλωσορίσω τους επισκέπτες μας που είναι πρώην δήμαρχοι από μια περιφέρεια στην Ιταλία Φριούλη, Βένετο, Βενετία και Τζούλη. Καλώς ορίσατε. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Ντεμόντε που είναι μέλος της Επιτροπής ε, Μεταφορών και Τουρισμού και ε, μέλος της Σοσιαλδημοκρατικής Ομάδας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και για τους χαιρετισμού από τους δημάρχους της περιοχής μου και εγώ ανταποκρίνομαι, ανταποδίδω το χαιρετισμό και μπαίνω στην παρέμβασή μου όχι για να θίξω τα ισχυρά σημεία που έχει ο τουρισμός, τα πλεονεκτήματα που μπορούν να ισχυροποιηθούν και στο μέλλον, διότι αυτό είναι δεδομένο. Θα ήθελα να υπογραμμίσω όμως αυτό που είναι σημαντικό για να διατηρηθεί η Ευρώπη σαν πρώτος προορισμός σε παγκόσμιο επίπεδο. Σίγουρα η τάση του τουρισμού είναι θετική, αυτό το γνωρίζουμε, αλλά θα πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε ότι αυτό εν μέρει οφείλεται και στον αντίκτυπο που έχει η κάποια αστάθεια στη Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή. Γι' αυτό θα πρέπει να επαγρυπνούμε, διότι δεν υπάρχουν μόνο αυτά τα προβλήματα, αλλά υπάρχουν και άλλοι στόχοι που είναι ανταγωνιστικοί εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλοι προορισμοί, χάρη σε άλλους παράγοντες όπως είναι η τιμή. Για να διατηρήσουμε την πρώτη θέση θα πρέπει να προωθήσουμε και τις πιο απόμακρες περιοχές, τις λιγότερο γνωστές, όπου είναι όμως πραγματικά κοσμήματα. Και εκεί ανήκουν μικρές πόλεις, ιστορικές τοποθεσίες ε, και μικρά χωριά ορεινά. Αλλά για να μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί στην πρόθεση και διαφήμιση πρέπει να βασιστούμε στα, στην πληροφορική μέσο. Σίγουρα είναι απαραίτητο να προσφύγουμε στην ψηφιοποίηση στο πεδίο του τουρισμού. Συνεπώς να γνωστοποιήσουμε στους πολλούς και στις απόμακρες ε, αγορές ε, τους πιο απόμακρους προορισμούς. Μέσα είναι και η εικονική και αυξημένη πραγματικότητα, διότι θέλει ο καταναλωτής όχι μόνο να προγραμματίσει το ταξίδι του, αλλά θέλει να έχει και μία εμπειρία ε, ίδια. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ε, τις διάφορες πλατφόρμες που υπάρχουν, διάλεξε ριζικά ο κόσμος ταξιδιού. Ε, και έτσι θα δημιουργηθούν, ε, θα έχουμε και νέους τουρίστες, προσελκύσουμε. Για να το κάνουμε αυτό πρέπει να δημιουργήσουμε τις αναγκαίες δεξιότητες, γνώση, να επενδύσουμε επί της εκπαίδευσης στοχευμένης, δηλαδή να μιλούνται περισσότερο οι ξένες γλώσσες, περισσότερες ξένες γλώσσες. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να προσεγγίσουμε άλλες ε, κουλτούρες και διαφορετικές ευαισθησίες. Ουσιαστικά θα πρέπει να βασιστούμε περισσότερο στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Πολύ συχνά το λέμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι πρέπει να ευνοήσουμε για την εποχικότητα, να, όλο το χρόνο υπάρχει ο τουρισμός και έτσι να εκμεταλλευτούμε περισσότερο τους προορισμούς που τώρα ε, τους δέχονται επισκέπτες μόνο με εποχή του χρόνου. Λοιπόν, τόποι που έχουν μεγάλη δυνατότητα υποδοχής θα πρέπει να γίνουν ελκυστικοί κυρίως ε, με διάφορα συνέδρια, ε, συνελεύσεις και ε, τον τουρισμό αυτών. Θα πρέπει να μείνουμε και εκτός συνόρων δραστήριοι σαν Ευρώπη. Ε, θα πρέπει να αρθούν τα διάφορα εμπόδια που υπάρχουν. Τα εμπόδια ποια είναι. Οι θεωρήσεις, θεωριστικές βίζες που χρειάζονται αναφέρομαι, τώρα μιλήσαμε και στις προηγούμενες παρεμβάσεις γι' αυτό, για χώρες όπως η Κίνα, που είναι μια βάση αναδυόμενη τουρισμού με την απλούστευση τη χορηγήσεω θεωρήσεων. Υπολογίστηκε ότι μόνο λαμβάνοντα υπόψη την Κίνα, την Ινδία, τη Ρωσία, τη Σαουδική Αραβία και την Νότια Αφρική και την Ουκρανία, θα αυξανόταν ο πληθυσμό προ το χώρο Σέγγεν κατά 130 δισεκατομμύρια ευρώ σε 5 χρόνια. Μία αύξηση 1,3 εκατομμύρια θέσεων εργασία θα οδηγήσει αυτή η αύξηση. Άλλη πτυχή αφορά την επιτροπή στην οποία ανήκω, δηλαδή μεταφορών και τουρισμού. Διότι οι δύο πτυχέ είναι αλληλένδετε στενά. Δεν υπάρχει ένα προορισμό αν δεν είναι δυνατόν να φτάσει κανεί εκεί. Δεν υπάρχει ένα προορισμό όχι μόνο που μπορεί να πάει κανεί, αλλά και να είναι προσβάσιμο εύκολα. Αυτό που πρέπει να επαναληφθεί είναι ότι θα πρέπει να προωθήσουμε έναν τουρισμό για όλου. Ε, κλείνω, Πρόεδρε, λέγοντα ότι εκτιμώ πάρα πολύ αυτή την πρωτοβουλία τη σημερινή, διότι θα πρέπει αυτή να είναι, να είναι ένα ραντεβού που θα πρέπει να επαναληφθεί. Διότι μόνο μέσω μια ε, ομαδική ισχυρή συνεργασία μπορούμε να πετύχουμε η Ευρώπη να διατηρηθεί στην πρώτη θέση σαν προορισμό σε παγκόσμιο επίπεδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ντεμόντε και με χαρά τώρα θα δώσω το λόγο σε άλλη συνάδελφο της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, την κυρία Μπιλμπάου Μπαραντίκα, από τη χώρα των Βάσκων και την ομάδα των Φιλελευθέρων. Κυρία Μπιλμπάου, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους επισκέπτες. Όπως είπαμε, χρειαζόμαστε κάποιες πολιτικές έτσι ώστε να έχουμε ανταγωνιστικό, ποιοτικό τουρισμό. Κατά αναλογία αυτό είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, η ισχύ μας είναι ότι έχουμε κάνει την ποικιλομορφία μας ένα στοιχείο συμβίωσης και ε, δημιουργίας πλούτου. Αυτό θα πρέπει να βοηθήσουμε ανάπτυξη να είναι βιώσιμη και να βασίζεται στη γνώση αλλά χωρίς αποκλεισμούς. Ευρώπη, τουρισμός ποιότητα. Αυτό είναι. Έχουμε μια ε, ποιότητα και μια ποικιλομορφία γλωσσική, πολιτισμική και αξίζει τον κόπο να τη ζήσει κανείς. Μια ε, εμπειρία ε, μοναδική. Γιατί όποια γεύση και να διαλέξει κανείς, η μάρκα Ευρώπη σημαίνει υψηλή ποιότητα. Εγώ είμαι από τη χώρα των Βάσκων και την εκπροσωπώ εδώ. Είναι μια γωνιά της γης που έχει μια παλιά πανάρχια γλώσσα και μια ε, ε, καταπληκτική φυσική ομορφιά και κληρονομιά. Και θέλουμε να τη μοιραστούμε με τους άλλους είναι μια προσφορά μας σε μια αγορά όλο και πιο ανταγωνιστική. Το 2016 κλείσαμε με αύξηση κατά 9,8% του αριθμού των τουριστών που επισκέφτηκαν τη χώρα των Βάσκων και 12% αυξήθηκαν οι ε, διανυκτερεύσεις. Εδώ και 10 χρόνια είναι αυξητική αυτή η τάση ε, σε ένα γενικότερο πλαίσιο που δεν δείχνει την ίδια αύξηση. Οι κάτοικοι είναι λίγοι, κάτω από 2 εκατομμύρια και έχουμε 1.500 επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 90.000 πρόσωπα και αυτό βοηθάει για τη σταθερότητα. Όπως γνωρίζετε το 2011 ε, ξεπεράσαμε ε, μια εποχή βίας που μας εμπόδιζε να αναπτυχθούμε. Ε, και έτσι έχουμε επιτύχει την αηφορία, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα έκτοτε. Και προσπαθούμε να δώσουμε ε, ένα τρόπο ζωής, ε, ανεπανάληπτους τόπους και τρόπους ζωής ε, που δεν υπάρχουν πουθενά άλλου. Έχουμε πραγματικά αντικειμενικές συνθήκες που αξίζει τον κόπο να απολαύσετε. Αλλά χρειάζεται ακόμα τεράστια προσπάθεια προβολής μέσω του Μουσείου Guggenheim που είναι εμβληματική προσφορά ή ας πούμε ο καθεδρικός ναός στη Βιτόρια Γαστέης. Θα πρέπει τις αξίες μας αυτές να τις μεταφράσουμε σε τουριστική ε, αξία. Με δέκα ε, ενέργειες κλειδιά προσπαθούμε να βελτιώσουμε τη θέση μας, το μερίδιο αγοράς μας και να μετρήσουμε την ανάπτυξή μας. Αυτοί είναι πυλώνες ενός σχεδίου που θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2020 και εμπνέεται από τις στρατηγικές του 2010 ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρώπη, πρώτος παγκόσμιος ε, τουρισμός και το 2014 για τον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό. Θα πρέπει να διδαχθούμε από τις επιτυχίες και τις αποτυχίες μας να ε, διαφυλάξουμε αυτό που περιμένουν να βρουν οι επισκέπτες, μια μοναδική ανεπανάληπτη ποιότητα που είναι φτιαγμένη από γεύσεις, από τη γαστρονομία μας, ε, που έχουμε ε, ανακάτοικο τα περισσότερα στέρια μισελέ στην Ευρώπη. Και έχουμε ε, το τσακολί, το κρασί μας, επίσης ανεπανάληπτο ή κάποια κρασιά από τη Ριόχα. Έχουμε φεστιβάλ jazz, φεστιβάλ κινηματογράφου στο Σαν Σεμπαστιάν. Αυτό δεν είναι υψηλή ποιότητα για την Ευρώπη σε όλο τον κόσμο. Ε, μια χώρα, μια περιφέρεια που είναι αστέρι, μισελέν. Δεν θέλουμε να πεθάνουμε όμως από την επιτυχία μας. Το Σαν Χουάν Γαστελγουάτσε είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Είναι μοναδικό ε, αυτό το τοπίο και υποψήφιο για το καλύτερο κινηματογραφικό σκηνικό στην Ευρώπη. Πώς θα διαχειριστεί κανείς αυτή την επιτυχία. Είναι η βιωσιμότητα το κλειδί πιστεύουμε για να έχουμε ακριβώς την ποιότητα που ε, απαιτεί το παγκόσμιο κύρος. Δεν μου μένει παρά να σας καλέσω να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία που αξίζει τον κόπο στη χώρα των Πάσκων. Ευχαριστώ. Vielen herzlichen Dank. Σας ευχαριστώ θερμά. Θα δώσουμε τώρα το λόγο σε έναν άλλο συνάδελφο από το Κοινοβούλιο, από την Κροατία. Και νομίζω πως ε, ε και η Κροατία ε, κατάφερε να προσελκύσει πολλούς οπαδούς του Game of Thrones, ειδικότερα μετά από τις ε, που έγιναν στον Τουμπρόβνικ τουλάχιστον. Καλωσορίζω λοιπόν θερμά τον ε, συνάδελφο ε, ο οποίος είναι ε, μέλος της Επιτροπής για την Περιφερειακή Ανάπτυξη και από την πολιτική ομάδα των Νέων Φιλελεύθερων. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Γεννήθηκα στο Πόρετς. Και γιατί το λέω αυτό που γεννήθηκα. Διότι το Πόρετς είναι η Μητρόπολη του κρατικού τουρισμού, διότι η Ίστρια είναι η περιοχή για την οποία, είχα τα, την οποία εκπροσωπούσα επί 12 χρόνια. Είναι πολύ τουριστική περιοχή στην Κροατία, πάνω από 50% του τζίρου του τουρισμού της Κροατίας ε, παράγεται εκεί. Είναι πολύ ελκυστική περιοχή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε ευρύτερο πλαίσιο. Η Κροατία είναι πολύ της μόδας. Και η Ίστρια είναι in. Αυτό ισχύει και για άλλους προορισμούς, όχι μόνο στην Ίστρια αλλά και σε άλλες περιοχές της Κροατίας. Εργάστηκα ε, και σε ξενοδοχείο μετέφερα βαλίτσες έγινα και υπουργό τουρισμού της Κροατίας. Με κάλεσε να αναλάβω τη θέση αυτή ο Κροάτης Πρωθυπουργό. Στο τέλος, όμως, έγινα, έγινα υπουργό Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και όχι τουρισμού. Ο τουρισμός είναι πάρα πολύ σημαντικός για όλους μας στην Κροατία. Και είναι σημαντικό για όλους μας που είμαστε πολιτικοί να έχουμε κάποια εμπειρία από τον τουρισμό. Η πιο σημαντική μου εμπειρία ήταν όταν έγινα νομάρχης στην Ίστρια. Το 2002 ετοιμάσαμε ένα σχέδιο για τον τουρισμό, για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή της Ίστρια. Συνεργαστήκαμε με άλλη περιοχή στην κατάρτιση του σχεδίου, με την Καταλωνία και θέλαμε να αποφύγουμε τα σφάλματα της Καταλωνίας. Και έτσι ξεκινήσαμε πάνω από 300 άνθρωποι ενεπλάκησαν στη σύνταξη του σχεδίου αυτού. Η επιτυχία μας στον τουριστικό τομέα δεν ήταν τυχαία, εργαστήκαμε σκληρά γι' αυτό. Τώρα, όλοι οι ομιλητές σας κάλεσαν να, έρθετε στην περιοχή τους και εγώ το ίδιο θα κάνω. Σας επευθύνω πρόσκληση. Αυτή είναι η δική μου εμπειρία για την περιοχή μου, για την Ίστρια. Δράτω με της ευκαιρίας να πω το εξής. Θα ήθελα να ξεκινήσω κάτι το οποίο επεξεργαζόμουν τελευταία τρία ετία. Νομίζω ότι αυτή η εκδήλωση υψηλού επίπεδου είναι το κατάλληλο σημείο και ο χώρο. Ακούσαμε σωστά επιχειρήματα του κυρίου Ταγιάννη. Έξοχη ομιλία του κυρίου Ταγιάννη. Χρειαζόμαστε Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τον Τουρισμό. Πρέπει να χειριστούμε, να διαχειριστούμε τον τουρισμό. Αν θέλουμε να παραμείνουμε στην πρώτη θέση, σαν τουριστικός προορισμός, χρειαζόμαστε αυτό το φορέα, αυτό τον οργανισμό. Έχουμε δωδεκάδες άλλες τέτοιες οργα... Ε, οργανώσεις, οργανισμούς. 10% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ ε, είναι ο τουρισμός, απασχολεί πάνω από 10 εκατομμύρια ανθρώπους. Ταυτόχρονα δεν έχουμε το θάρρος να πούμε ότι χρειαζόμαστε άλλη μια ευρωπαϊκή υπηρεσία, άλλον έναν ευρωπαϊκό οργανισμό. Ίσως άλλοι οργανισμοί να μην χρειάζονται, αλλά όχι αυτός. Αυτόν τον χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε συντονισμό όσον αφορά τις δραστηριότητε του τουρισμού. Να βοηθήσει ε, στην ανταλλαγή εμπειριών, να θεσπίσει και να προωθήσει καινοτομία. Και αυτό πρέπει να γίνει προ όφελο όλων των αναμειγνιωμένων στον τουρισμό. Θα παραμείνει ο ανταγωνισμό, αλλά χρειαζόμαστε ένα κοινό φορέα. Και γι' αυτό καλό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει τη δημιουργία αυτού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τουρισμού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο σε κάποιο προσκεκλημένο, γιατί θα πρέπει να φύγει να πάει στο Μιλάνο, αλλιώς θα χάσει την πτήση του. Είναι ο κύριος Μπρατσίνη, πληρωτής πρόεδρος ε, του Ιδρύματος Αλτα Γκάμα, ε, που εκπροσωπεί πολυτελείς ε, επιχειρήσεις από την Ιταλία και επίσης συνεργάζεται σε μια συμμαχία για τη δημιουργική βιομηχανία. Καλώς ορίσατε κύριε Βρόντσιν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, εκπροσωπώ περισσότερο τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό και όχι τον Ιταλικό. 500 εταιρείε ευρωπαϊκές τουρισμού υψηλού επίπεδου ενώθηκαν. Έχουν στα χέρια τους 70% μερίδιο της παγκοσμίου αγοράς. Ο τομέας μας είναι από τους ελάχιστους στους οποίους η Ευρώπη έχει τόσο μεγάλο, απίστευτο ποσοστό και επιτυχία. Άρα, αναφυσβήτητα, η αξία ε, το αφορολόγητο, τους αγοράς στην Ευρώπη ήταν περίπου 40 ε, δις το 2016 και το τρέχον έτος πρέπει να φτάσουμε 45 δις ευρώ. Πριν από τρία χρόνια μια έρευνα του ΟΗΕ έδειξε ότι κατά μέσο όρο οι επισκέπτες στην Ευρώπη αγοράζουν ε, προϊόντα πολυτελείας. Πάνω από 30% των κινήτρων επίσκεψης είναι η αγορά ε, πολύτιμων ε, αγαθών. Αγαθών πολυτελείας. Πάμε τώρα στο θέμα μας. Πώς να προωθήσουμε περαιτέρω την Ευρώπη ως τουριστικό προορισμό. Να είναι υπαριθμόν ένα προορισμός. Ακούσαμε κάποια πράγματα. Η διευκόλυνση των ταξιδιωτικών θεωρήσεων είναι σημαντικότατη. Έχουμε την ψηφιακή επικοινωνία, σημαντική πρόκληση για πολλές περιοχές και για υπέροχες πόλεις και περιβάλλοντα ευρωπαϊκά. Να σας επιστήσω την προσοχή σε κάτι. Είναι κάτι που θεωρώ κρίσιμη σημασία. Διότι υπάρχει συσχετισμός μεταξύ τουρισμού και αεροπορικών εταιριών. Πολύ στενή σχέση. Το βλέπουμε όλοι. Όχι μόνο φέτος ή πέρσι συμβαίνει αυτό. Ότι υποφέρει ο τομέας πολυτελείας στην Ευρώπη πολύ τα τελευταία δύο-τρία χρόνια. Αν κατά μέσο όρο θεωρήσετε ότι έχουμε μία, δύο από τις εκατό αεροπορικές εταιρείες που έχουν θετικό ισοζύγιο βλέπουμε ότι δεν έχουμε μελλοντικέ προοπτικές στην Ευρώπη σε αυτό το τομέα. Όπως είπε η Επιτροπή Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μέλη του, της Επιτροπής Τουρισμού και Μεταφορών και εγώ τονίζω το ρόλο των μεταφορών και των νέων πολιτικών μεταφορών. Πόσο μπορούν να βοηθήσουν τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες να ανακάμψουν. Και αυτό θα οδηγήσει σε ανάκαμψη της αγοράς αγαθών πολυτελείας στην Ευρώπη. Κάτι που θα είναι πολύτιμο στον αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ. vielen, σας ευχαριστώ ε, θερμά κύριε Μπραντσίνη. Ε, καλή επιστροφή στο Μιλάνο. Ε, σας ευχαριστώ ότι πάλι που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας για την παρέμβασή σας. Περνάμε τώρα. Ή κανονικά θα έπρεπε να περάσουμε στον κύριο Κορσίνη, αλλά δυστυχώς ασθένησε ο κύριος Κορσίνη, που είναι ο αρμόδιος υπουργός τουρισμού από την περιφέρεια της Εμίλια Ρωμάνια αλλά η Λορένσα Μπαντάιο είναι εκείνη που θα τον αντικαταστήσει σήμερα εδώ, που είναι επικεφαλής του Περιφερειακού Γραφείου για την Εμιλία Ρωμάνια, εδώ με την αντιπροσωπεία δηλαδή τη ε, περιοχή αυτή στι Βρυξέλλε, οπότε τη δίνω κατευθείαν στο λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, διαβιβάζω του χαιρετισμού του Υπουργού μα, του κ. Κωσίνη, του Υπουργού Βιομηχανία. Ο κ. Κωσίνη δυστυχώ δεν μπορούσε να παραστεί. Η Εμίλια Ρωμάνια είναι ευγνώμων ε, έναντι του Πρόεδρου Ταγιάννη που απίφθηνε αυτή την πρόσκληση και που μας κάλεσε σε αυτή τη μοναδική εκδήλωση στρατηγικής σημασίας για όλους μας. Εν συντομία να μοιραστώ κάποια πράγματα μαζί σας. Πώς συμβάλλει η Εμίλια Ρωμάνια στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού τουρισμού και πώς ενισχύει την Ευρώπη στη θέση της που είναι υπαριθμόν ένα τουριστικός προορισμός, αυτό που συζητούμε μέχρι τώρα. Κάποια χαρακτηριστικά αρχικά. 2017 στοιχεία δείχνουν τον αντίκτυπο που έχει ο τουρισμός στις επενδύσεις και στις θέσεις απασχόλησης στην Εμίλια Ρωμάνια. Ο τουρισμός είναι στρατηγικός πυλώνας και κινητήρια δύναμη για την περιφερειακή οικονομία. Αριθμοί. 16 δις ευρώ ο τουρισμός αντιπροσωπεύει πάνω από το 11% του περιφερειακού ΕΠ. 44 εκατομμύρια παρουσίες που έχουν καταχωρηθεί ε, πριν από μερικές ημέρες μετά τον Αύγουστο. 9 εκατομμύρια φίξεις. Αυτά τα στοιχεία αυξάνονται. Όλα αυτά συμβάλλουν σε μείωση της ανεργίας που στην Εμίλια Ρωμάνια από 9 έπεσε στο 6,4% η ανεργία. Η Εμίλια Ρωμάνια είναι στην Ιταλία η τέταρτη πλέον τουριστική περιοχή της χώρας. Και όπως είπε ο κύριος Ντεμόντε, ο συγκητής, είναι πολύ προσβάσιμη η περιοχή. Σε πολύ καλή θέση. Τώρα, όπως τα βλέπουμε σε περιφερειακό επίπεδο, ποια εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν μέχρι τώρα από την Εμίλια Ρωμάνια. Πρώτα απ' όλα, η Εμίλια Ρωμάνια είναι νομοθετική. Μπορεί να νομοθετεί. Έχει περιφερειακό νομοθέτημα. Νόμο βασικό δικό της για τον τουρισμό. Και πιο συγκεκριμένα. Έχουμε βρει νέα εργατήλια προώθηση στην αγορά. Μάρκετι. Ε, εμπειρία μέσω της Εμίλια, Via Emilia Experience αποκαλείται. Εμπειρίες μέσω της κοιλάδας των φαγητών, ε, ε, ε αυτοκινήτων ε, και πάθους, αν θέλετε. Μέσω αυτών των διαδρομών, των τουριστικών, θέλουμε να αυξήσουμε τη διεθνοποίηση της προσέγγισης και την ταυτότητα της μάρκας, αν θέλετε. σε ευρωπαϊκό επίπεδο τώρα. Τι κάνουμε. Η Εμίλια Ρωμάνια στην Ευρώπη. Συμβάλλει σημαντικά με κάποια εργαλεία. Πρώτον, αποτελεσματική πραγματική συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, διαθωτικά ταμεία, στον ορίζοντα 2020 και στο κόσμο. Και και ο Γιάκοβιτς και γι' αυτό αναφέρω στη μακροπεριφέρεια Αδριατικής Ιωνίου, που είναι σημαντική διάσταση αυτή για τον τουρισμό. Δεύτερον, η Μίλια Ρωμάνια δραστηριοποιείται ιδιαίτερως στα σημαντικά ευρωπαϊκά δίκτυα. Ακούσαμε διάφορα να αναφέρονται. Διάφορα δίκτυα, όπως είναι του πολιτισμού και του τουρισμού, όπως το BRIC. Και σωστά ανέφερε το πολιτισμό η πρόεδρος. Ισορροπία μεταξύ πολιτισμού και τουρισμού. Τρίτον, καλωσορίζει η περιοχή μου το 2018 που είναι Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και θα είναι ενεργός εταίρος στην προσπάθεια η Εμίλια Ρωμάνια. Και το έτος Ευρωπαϊκής Ενώσεως Κίνας το καλωσορίζουμε. Οι αρμόδιες αρχές πάνε στο Χαντόγκ που είναι η περιοχή μας ε, με την οποία συνεργαζόμαστε τον Νοέμβριο. Για όλους αυτούς τους λόγους η Εμίλια Ρωμάνια υποστηρίζει ανανεωμένη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ενώσης για τον τουρισμό, όπως είπε και ο Υπουργός ο κ. Και είναι σε θέση να διαθέσει ειδικού πόρους στο νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και τα προγράμματα μετά το 2020 για αυτό το σκοπό. Και ελπίζουμε να υπάρχει ιδιαίτερο πρόγραμμα, ειδικό πρόγραμμα, ειδικό κονδύλι για τον τουρισμό. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τουρισμού, κύριε Γιάκοβιτς, κύριε Γιάκοβιτς, γιατί όχι. Ευχαριστούμε τον κύριο Ταγιάννη και σας κυρία Πρόεδρε για τις προσπάθειες αυτές, τις πολύ έγκαιρες για την οργάνωση αυτής της ε, διάσκεψης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ θερμά. Και για το διακρατιστή σας τα ισότερα σοβραχή πρόθεσμα, τον κύριο Κωσίνη, ε, περνάμε τώρα ε, σε μια επισκέπτρια που έρχεται και εκείνη από μακριά, που είναι ε, αναπληρώτρια ε, γενική διευθύντρια και οι γενικοί γραμματές του ε, Global Tourism Economy Forum όπου δίνεται βέβαια ιδιαίτερη έμφαση της τουριστικής ανάπτυξης σε σχέση με την Κίνα. Έχετε λοιπόν το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Επίτροπη, συμμετέχονται σήμερα εδώ. Με τιμή μου συμμετέχω σήμερα σε αυτήν την διάσκεψη ψηλού επίπεδου για τον τουρισμό. Και ε, θεωρώ πως ε, είναι ιδιαίτερα εύστοχο το γεγονός ε, ότι παρουσιάζω σήμερα εδώ αυτό το παγκόσμιο φόρμα για την τουριστική οικονομία που διοργανώνεται κάθε χρόνο στο Μακάο της Κίνας προκειμένου να προωθηθούν αυτοί ε, ε, προορισμοί και ειδικότερα ε, η, η Κίνα ως η κύρια χώρα από την οποία προέρχονται οι τουρίστες σήμερα στον κόσμο. Δηλαδή όλο ένα και περισσότερο γίνεται αντιληπτός ο ρόλος που μπορεί να παίξει ο τουρισμός σε ό,τι αφορά τον οικονομικό μετασχηματισμό, την ανάπτυξη αλλά και την πολιτιστική πρόοδο. Ε, ήδη ε, ε, η Κίνα έχει δημιουργήσει έναν ε, πυλώνα πολιτική σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα τον τουρισμό, που ταυτόχρονα συνοδεύεται αναπτυξιακή στρατηγική και δημόσια διπλωματία. Ο τουρισμός μάλιστα ενσαρκώνει και την πρωτοβουλία τη μία ζώνης ενός δρόμου με πρωτοβουλία του Προέδρου Xi Jinping, προκειμένου να προωθηθεί περισσότερο ο ανοιχτό χαρακτήρα στη συνεργασία και τα κοινά ωφέλη. Η επίσης χρησιμοποιεί τον τουρισμό για να συνδεθεί με τον κόσμο και να δημιουργήσει ευκαιρίες οι οποίες προέρχονται από την οικονομική της ανάπτυξη. Το 2012 ε, το φόρουμ αυτό, το GTEF, δημιουργήθηκε ως η πρώτη πρωτοβουλία δημοσίου και ιδιωτικού ε, τομέα σε συνεργασία με πολλέ ε, παγκόσμιε οργανώσει προκειμένου να προωθηθεί η δημιουργία ακριβώ ενό βιώσιμου παγκόσμιου τουρισμού. Με την Κίνα στον πυρήνα αυτή τη ε, πρωτοβουλία αφού η Κίνα εδώ παίζει το ρόλο ενό σημαντικού εταίρου. Οι συνέργειε αυτέ, οι διεθνεί συνέργειε του GTEF και συνεργασίες είναι για παράδειγμα ο WTO των Ηνωμένων Εθνών, η Συνομοσπονδία για την ε, για τα ταξίδια στην Κεντρική και Νότια Ασία ε, και ιδιαίτερα ε, με την τουριστική υπηρεσία του, την Κινέζικη Υπηρεσία Τουρισμού και ειδικότερα την υπηρεσία του Μακάο. Και αναδείχθηκε ιδιαίτερα περισσότερο όταν πέρσι αναφέρθηκε ως μία από τις 19 κύριες πρωτοβουλίες οι οποίες θα λάβουν υποστήριξη ειδικότερα στο Μακάο. ΚΑΟ επιλέχθηκε ως έδρα του φόρουμ αυτού γιατί με 450 ε, χρόνια αυτή της, ε, του παντρέματος αν του πολιτισμού μεταξύ Ανατολής και Δύσης έχει ένα ιδιαίτερο ρόλο και ε, λαμβάνει ένα μεγάλο μέρος των ε, ε τουριστών της Κίνας. Από τότε δηλαδή που επανεντάχθηκε στην Κίνα από 6 εκατομμύρια τότε έχει φτάσει στα 30 εκατομμύρια ε, τουρίστες με ένα ε, ε, πληθυσμό μόνο 600.000 και ο οποίος διαμένει σε 32 μόνο τετραγωνικά χιλιόμετρα. Και τώρα το GTF έχει ε, δεσμευτεί στο να δημιουργήσει περισσότερα ακόμα συνέργεια σε ό,τι αφορά διαφορετικέ περιφέρειε, δημόσιου και ιδιωτικού φορεί, αλλά και μεταξύ ανθρώπων, προκειμένου να υπάρχει περισσότερη ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών, προκειμένου να υπάρξουν καλύτερε αντιστοιχίε επιχειρηματικών ευκαιριών και καλύτερε συνεργασίε σε επιχειρησιακό επίπεδο. Από το 2012 το GTF έχει συμπεριλάβει 7.000 ε, συμμετέχοντες από 63 διαφορετικές χώρες και ε, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων περιφερειακών ε, οργάνων και διάφορους ε, πάρα πολύ ε, επιφανείς ομιλητές ε, με συνολική κάλυψη από τα μέσα που άντυξε την αξία των 30 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Κίνα έχει εδώ και πολύ καιρό αναγνωρίσει τη σημασία των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας και προωθεί ειδικότερα τον τουρισμό, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά την Πορτογαλία και την Ισπανία, αναδεικνώμε το 2013, το 2016 την Γαλλία και φέτος τις χώρες της Ανατολικής και της Ευρώπης. βασιζόμενοι σε αυτές τις σταθερές και διαρκεί ε, σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και Κίνα, ε, και λαμβάνοντα υπόψη αυτή τη βούληση για περαιτέρω συνεργασία, μπορώ να σας μέσω του GTEF να σας αναδείξω και την Κίνα ω έναν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα τουριστικό προορισμό. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ και ε, ελπίζω να σας δω όλους ε, του χρόνου στο Μακάο, κατά το επόμενο δηλαδή, την επόμενη συνεδρίαση του Φόρουμ το 2018. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ακολουθεί η, η κυρία Μπολιέ, που είναι πρόεδρος μιας εταιρείας που ασχολείται με ε, πολυτελείς κατοικίες στην Ευρώπη και στην Κίνα. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ε, πρωτοβουλία και αυτός ο συνδυασμός. Value Retail ονομάζεται η εταιρεία. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομη. Πριν από 21 χρόνια, decided... Αποφασίσαμε να αναπτύξουμε όχι προορισμούς, μάλλον όχι ένα εμπορικό κέντρο, αλλά προορισμούς. Δηλαδή το να δημιουργήσει ένα προορισμό χρειάζεται κάποια κριτήρια. Να έχει συνδέσεις. Εξαρτάται από το δημόσιο τομέα αυτό, δηλαδή να υποδομές, αεροδρόμια και ε, συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά για να έχουμε ε, πραγματικά τις διασυνδέσεις. Έχουμε δημιουργήσει δηλαδή εμπορικά κέντρα που είναι ε, προορισμοί για να πηγαίνει κανείς να ψωνίζει, outlets. Κάθε χωριό λοιπόν το οποίο ανοίξαμε και στο οποίο επενδύσαμε θα πρέπει να λέει μια ιστορία από μόνο του το ε, χωριό αυτό με τα καταστήματα για να προσελκύει τουρισμό. Στη συνέχεια θα έπρεπε όλα αυτά να τα διαδώσουμε αυτή την κοινότητα και αυτή την πολιτισμική οικονομία κάθε φορά. Άρα θα έπρεπε να ε, επενδύσουμε σε υψηλότερα προσόντα ε, και τουριστικούς διευθυντές και αυτή τη φορά ε, φέτος ε, απασχολούμε 70 διευθυντές τέτοιων ε, εμπορικών χωριών με καινοτομία. Άρα θα πρέπει να προχωρήσουμε στη ψηφιοποίηση. άλλη δέσμευση και στόχος μας. Άρα είμαστε πρωτοπόροι σε αυτή την κατηγορία τουρισμού και έχουμε 11 χωριά στην Κίνα και στην Ευρώπη με 37,4 ε, εκατομμύρια ε, τουρίστες και με αύξηση 10% στις πωλήσει. Με τάσεις αντίστοιχες να αναμένουμε για φέτος. Αυτή όμως η ε, επιτυχία δεν νοείται χωρίς τη στενή συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Είμαστε μέλη του WTTC, του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού. Και θα συνεχίσουμε να προωθούμε αυτές τις δράσεις και τη Λευκή Βίβλο. Για το τι σημαίνει ο αγοραστικός τουρισμός για μια πόλη, για ε, την περιοχή και τι αντίκτυπο έχει σε αυτή. Στην Ισπανία ε, συνεργαζόμαστε με την κυβέρνηση της Καταλωνίας. Και σύντομα καταφέραμε να μετρήσουμε τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει για τα, ωράρια των καταστημάτων, των εμπορικών, για την εργασία ε, την Κυριακή. Επιτύχαμε μεγαλύτερα ωράρια να ανοίγουν τα καταστήματα τις Κυριακές με άμεση επίπτωση 20% αύξηση στην απασχόληση και 20% αύξηση στις πολίτες και στην Βαρκελόνη είναι ανοιχτά 7 μέρες την εβδομάδα ε, τα καταστήματα για τουρίστες, είτε αυτοί είναι ε, από την ίδια τη χώρα, ε, από το εξωτερικό, από την Ευρώπη ή διεθνής. Κοινή λοιπόν προσέγγιση και συναντήληψη χρειάζεται του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα για να πετύχει οτιδήποτε τέτοιο εγχείρημα. Είτε πρόκειται για την ασφάλεια στα σύνορα, είτε ε, για τις θεωρήσεις διαβατηρίων, ενώ εξασφαλίζεται ελεύθερη κυκλοφορία. Ε, αυτός είναι ένας στόχος που ελπίζουμε να επιτύχουμε σε πολύ στενή συνεργασία με το δημόσιο τομέα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Βόλιε. Και τώρα ερχόμαστε στον Εντράδο Σανταντέρ, αν το λέω καλά, ε, Διευθύνων Σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, Τουρισμού, ε, ταξιδίων μάλλον. Κοιτάξτε, Ευχαριστώ τον πρόεδρο, τον κύριο Ταγιάννη, διοργάνωση τη διάσκεψη και όλα τα κόμματα του Κοινοβουλίου. Έγινε πολλή δουλειά αυτή η διάσκεψη. Δούλεψαν πολλοί υπάλληλοι και, και πολλά προβλήματα. Δεν τα βλέπουμε αυτά, αλλά έχουν λυθεί τα προβλήματα και συγχαρητήρια για τη διάσκεψη και χαρούμενη ημέρα τουρισμού εύχομαι σε όλους. Εκπροσωπώ σήμερα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδίων. Είναι αρκετά παλιός φορέας, ιδρυθήκαμε το 1948. Είμαστε πιο παλιοί από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση των πραγμάτων. Και είναι ηρωνική ιστορία. Όταν ιδρύθηκε ο οργανισμός μας, υπήρχαν κάποιοι που θεωρούσαν ότι ο τουρισμός θα μπορούσε να είναι ο κινητήρας κινητήρια δύναμη της οικονομίας ευρωπαϊκής και της ανάπτυξης μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τώρα μετά από 70 χρόνια δεν μιλάμε για τίποτα άλλο. Ο τουρισμός ήταν και είναι η κινητήρια δύναμη για ανάπτυξη. Δεν το φανταζόταν παλιά μάλλον και το φαντάζεται ο κόσμος τώρα. Ε, εκπροσωπούμε 33 ε, οργανισμούς τουρισμού της Ευρώπης. Εργαζόμαστε στο μάρκετινγκ, διεκδικούμε την ελευθερία ταξιδιών, διευκόλυνση, διευκόλυνση των ταξιδιών διεκδικούμε, βιώσιμο τουρισμό επιδιώκουμε και πολεμάμε γι' αυτό και πολεμάμε και για διασυνδεσιμότητα. Πρέπει να συνδέονται οι τόποι της Ευρώπης, όχι μόνο εσωτερικά αλλά και με την τρίτη αγορά. Μετά, άλλος τομέα στον οποίο κινούμεθα και είμαι περήφανος γι' αυτό διότι με διάφορους φορείς, ε, Διεθνή Συνομοσπονδία Τουριστικών ε, Οργανισμών και με το Μακάο, με όλους αυτούς κάνουμε έρευνα. Να σας δώσω κάποια στοιχεία όσον αφορά την έρευνα. Τι γίνεται στην Ήπειρο όμως στον τουρισμό. Η Ευρώπη είναι από τους καλύτερους προορισμούς ταξιδίων στον κόσμο. Το 2016 είχαμε ανάπτυξη για τον τουρισμό. Εντυπωσιακή ανάπτυξη του τουρισμού παρά τα οικονομικά και πολιτικά προβλήματα και παρά τα προβλήματα ασφαλείας. Πάνω από 50% του μεριδίου του τουρισμού στην αγορά έχει η ε, Ευρώπη. Πάνω από 630 εκατομμύρια αφήξεις τουριστών είχαμε στην Ευρώπη το 2015. Μας λένε ότι χάνουμε μερίδι της αγοράς. Αλλά δεν είναι και τόσο μεγάλο πρόβλημα θα έλεγα. Το θέμα είναι να μην χάνουμε ανταγωνιστικότητα. Αυτό είναι το πρόβλημα που έχει η Ευρώπη όπως είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τουρισμού, αρκετοί προορισμοί ε, τουριστικοί αναπτύχθηκαν τελευταία. Η Νότια Ευρώπη εξακολουθεί να προσελκύει τους περισσότερους τουρίστες και μετά έρχεται η Δυτική Ευρώπη. Η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη την χάνουν μεγαλύτερης προσοχής και γιατί θεωρούνται και ασφαλείς προορισμοί αυτές, αυτοί οι προορισμοί για το έτος Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Κίνας. Πρέπει να γίνει μνήα της Κίνας. Η αγορά της Κίνας δείχνει κάποια ανάπτυξη με μέτρους ρυθμούς και προπτικές θετικές φαίνονταν το 2016. Πέρσι είχαμε 10 εκατομμύριο αφήξεις από την αγορά και αυξάνεται τα τελευταία πέντε χρόνια συνεχώς ο αριθμός επισκεπτών από την Κίνα. Προσελκύει περίπου 12% κάθε χρόνο της κινέζικης αγοράς η Ευρώπη. Υπάρχει μεγάλη δυνατότητα αύξησης αφήξεων από την κινέζικη αγορά. Περιφερειακές τάσεις στην Ευρώπη. Ε, ε, Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο ε, οδηγούν στην ανάπτυξη του τουρισμού εντός Ευρώπης και παραμένουν περιοχές που δίνουν θετικές προοπτικές είναι σταθερέ οι οικονομικές καταστάσεις, η οικονομική κατάσταση στην Ευρωζώνη. Όμως υπάρχουν προβληματισμοί για την ασφάλεια και ίσως τότε οι ταξιδιώτες να πηγαίνουν αλλού και ίσως θα μπορούμε να καταπολεμήσουμε και τον εποχιακό χαρακτήρα του τουρισμού. Υπάρχει τουρισμός όλο τον χρόνο υπάρχουν προβληματισμοί για λόγους πολιτικούς και ασφαλείας, αλλά εξακολουθεί να είναι ελκυστική η Ευρώπη για τουριστικός προορισμός. Για να παραμείνει η θέση μας πρώτη στον κόσμο, η ψήφιση σημασία είναι να παραδεχτούμε την ανάγκη να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί. Σε ένα τομέα που προσαρμόζεται γρήγορα ε, ο τομέας αυτό και από τις παραδοσιακές αγορές και από τις αναδυόμενες επηρεάζεται πρέπει να προσέξουμε την απόρρια ανταγωνιστικότητα. Εκεί πάντα, πάντα υπάρχει λύση, η συνεργασία. Είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Και αν θέλουμε να είναι υπαριθμόν ένα η Ευρώπη στον τουρισμό, θα πρέπει να μάθουμε να συνεργαζόμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά. Ε, κύριε Σανταντέρ. Ε, και, εγώ, ε, και να περάσουμε τώρα στον κύριο Ζαουλού που έχει έρθει και εκείνο από μακριά ε, που είναι ολοκληρωτός εκτελεστικός διευθυντής σε ό,τι αφορά τις στατικές και επενδυτικές σχέσεις της ΖΕΤΡΙΠ, η οποία είναι ένα ταξιδιωτικό γραφείο. Ε, παρακαλώ, έχετε το λόγο κύριε Ζαουλού. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας και σας Πρόεδρε για αυτή τη διάσκεψη υψηλού επίπεδου που μας προσκαλέσατε. Είμαστε ε, το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό γραφείο στον κόσμο ε, σε ό,τι αφορά την κίνηση και το δεύτερο ε, από εισπράξεις. Πάνω από δύο εκατομμύρια δωμάτια για την εκτρέψη έχουμε κλείσει και εκατομμύρια αεροπορικά εισιτήρια. Πάνω από 50 των Κινέζων που, 100 ε, ε, που ε, ταξιδεύουν χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας. Θα ήθελα να σας δώσω κάποια στοιχεία και αριθμούς που έχουμε για τους Κινέζους τουρίστες και κάποιες σκέψεις και προτάσεις που έχουμε για το πώς μπορεί να προωθηθεί ο τουρισμός στην Ευρώπη από τη σκοπιά της Κίνας και του κλάδου. Το 2016 είχαμε πάνω από 40 εκατομμύρια Κινέζους τουρίστες σε ξένες χώρες από την υπηρετική Κίνα που ε, ταξίδεψαν εκτός Κίνας, Μακάο, Ιβαν και Χονγκ Κονγκ. Από τα 40 εκατομμύρια, τα 20 πήγαν σε ασιατικές χώρες, Μαλαισία, Σιγκαπούρη, ε, Ιαπωνία και λιγότερη Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Ευρώπη. 10% του μεριδίου ε, αγοράς ε, των Κινέζων αστών πηγαίνουν στην Ευρώπη. 0,3% μόλις του κινέζικου πληθυσμού. Στι Ηνωμένε Πολιτείε πέρσι ήταν πάνω από 14 εκατομμύρια οι Αμερικανοί που επισκέφτηκαν την Ευρώπη. Υπάρχει πολύ μεγάλο δυναμικό για ανάπτυξη. Τα επόμενα 20 χρόνια μπορεί να τριπλασιαστεί έω να πενταπλασιαστεί ο αριθμός των Κινέζων τουριστών που επισκέπτονται την Ευρώπη. Για το 2016 πιστεύουμε ότι υπάρχουν δύο λόγοι ε, που οδήγησαν στην ε, χαμηλή προσέλευση των Κινέζων ήταν ότι το Γουάν ήταν πολύ χαμηλό στην ισοτιμία σε σχέση με το ευρώ, ακριβό το ευρώ. Οπότε ε, δεν ήταν πολύ εύκολο. Και δεύτερον, ο κόσμος άρχισε να εξερευνεί και, άλλες, ε, και άλλους προορισμούς, Ανατολική Ευρώπη, σκανδιναβικές χώρες και στην Ισπανία επίσης. Έχει διαφοροποιηθεί ο προορισμός Ευρώπη. Επίσης, ε, κατά μέσο όρο μένουν 10 μέρες οι Κινέζοι στην Ευρώπη, επισκέπτονται διάφορες χώρες, διάφορες πόλεις, στο ίδιο ταξίδι. Άρα αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον στοιχείο και πάντα η Γαλλία, η Ιταλία και η Ελβετία ε, είναι προορισμοί ε, τους οποίους επισκέπτονται μαζί σε ένα τουρ οι τουρίστες. Και επίση είναι πολύ μακριά εκεί, είναι μακρύ το ταξίδι και υπάρχει και ε, πρόβλημα στην Οπότε ο κόσμος προτιμά τα ομαδικά ταξίδια, τα οργανωμένα σε εκδρομές και όχι τα μεμονωμένα. Εάν θέλετε λοιπόν να προσελκύσετε περισσότερους τουρίστες, χρειάζεται ε, ε, συνεργασία μεγαλύτερη μεταξύ κρατών και πόλεων. Οι Κινέζοι τουρίστες ε, είναι συνηθισμένοι το κινέζικο σύστημα μεταφορών και εσείς ε, με τα τρένα και εδώ έχετε ένα σιδηροδρομικό δίκτυο πολύ ε, ανεπτυγμένο που μπορείτε να φαίνετε Κινέζους τουρίστες που να μην πηγαίνουν μόνο ε, σε προβεβλημένους προορισμούς αλλά και σε άλλους που συνδέονται με το τρένο. Επίσης Πολλοί από τους Κινέζους που έρχονται εδώ ταξιδεύουν για πρώτη φορά εκτός της χώρας τους και θα πρέπει να προωθήσουμε στην Κίνα, σε διάφορες πόλεις, όχι μόνο στο Πεκίνο και στη Σανχάη ε, και σε μικρότερες πόλεις, ε, άλλες ευρωπαϊκές πόλεις εκτός από τις πιο προβεβλημένες. Υπάρχουν και στις μικρές, μικρότερες κινέζικες πόλεις ε, δυνατότητες και με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούμε να σας βοηθήσουμε κι εμείς Ε, με ε, συνοδού στα σύνορα και στα τελωνία που να μιλούν κινέζικα με διευκολύνσεις θεωρήσεις, με αναγνώριση των διπλωμάτων οδήγησης και τέτοια άλλα πρακτικά βήματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και Τελευταία μας ομιλήτρια είναι η κυρία Κάστρο που είναι η διευθύντρια σε ό,τι αφορά ζητήματα ε, του τουρισμού ε, από την ε, περιοχή της Γαλλικίας στην πολιτική Ευχαριστώ πολύ και πολύ καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε για το μέλλον του τουρισμού που είναι τόσο σημαντικό για την οικονομία των χωρών μας και της Ευρώπης στο σύνολό της. Είναι ένας κλάδος γεμάτος προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες που και στην Ισπανία αλλά και στη Γαλλικία σημαίνει 11% του ΑΕΠ και 13% και 12% αντίστοιχα ε, της απασχόλησης. Εγώ εκπροσωπώ τη Γαλλικία, στο βορειοδυτική Ισπανία, συνορεύει με την Πορτογαλία, πάνω από 2.700.000 κατοίκους έχουμε, παρόλα αυτά πέρσι ε, υποδεχτήκαμε πάνω από 5.000.000 εκατομμύρια τουρίστες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το νούμερο, αλλά βεβαίως χωράει βελτίωση. Και μιλάμε πάντα για μια ανάπτυξη βιώσιμη. Είναι πάρα πολύ πλούσιο το τοπίο, ε, ο πολιτισμός και ε, φιλόξενη περιφέρεια. Πάνω από 1200 χρόνια, χάρη στο δρόμο του ε, Αγίου Ιακώβου της Κομποστέλα. Και ξέρετε ότι και ο Γκέτε έχει φτάσει, έχει κάνει το δρόμο αυτό μέχρι τον Άγιο Ιάκωβο της Κομποστέλα. Είναι πάρα πολύ προβεβλημένος διεθνώς αυτός ο δρόμος. Και τι είχε πει ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο δεύτερος από το Σαντιάγο της Κομποστέλα. Έλα εδώ να ανακαλύψεις τον εαυτό σου, να ανακαλύψεις ε, τις ε, ρίζες σου και... Ε, να αποκτήσει σε ψυχική ανάταση. Έρχονται από όλο τον κόσμο περιηγητές, προσκυνητές, ε, από 175 χώρες έχουμε προσκυνητές ε, και τάση αυξανόμενη χρόνο με το χρόνο. Πάνω από 300 ενώσεις και σωματεία υπάρχουν στον κόσμο, πάνω από 80.000 ε, άνθρωποι μιλούν για αυτή τη διαδρομή, το μονοπάτι του Αγίου Ιακώβου που είναι συνώνυμο της ομόνιας, της συμφιλίωσης, της αναγνώρισης, της φιλίας και το Συμβούλιο της Ευρώπης 23 Οκτωβρίου πριν από 30 χρόνια χαρακτήρισε ως ε, πρώτο ε, ταξιδιωτικό δρόμο και διαδρομή αυτή του Αγίου Ιακώβου, το προσκύνημα του Αγίου Ιακώβου στην Κοποστέλα και εργαζόμαστε για να το διατηρήσουμε θα πρέπει να συνεχιστεί αυτό το προσκύνημα ε, με τρόπο βιώσιμο. Γι' αυτό σχεδιάζουμε κάθε βήμα που κάνουμε ε, με ένα φύλλο πορείας, με έναν οδικό χάρτη για να αναπτύσσεται ε, βιώσιμα αυτό. Το 2021 είναι το επόμενο ιερό έτος. Αυτό το προσκύνημα χωράει ακόμα μεγάλη βελτίωση και ο δρόμος περνάει πάνω ε, από 100 κοινότητες από τις 313 που έχουμε ε, στη Γαλλικία. Η περιφέρειά μας επίσης είναι ε, παράκτια 1.600 χιλιόμετρα ακτών. Έχουμε 16 ε, ρίας που είναι κάτι φιόρδ που μπαίνουν γλώσσες της θάλασσας μέσα ε, στη γη με πολύ πλούσια ε, χλωρίδα πανίδα με επαγγέλματα ναυτικά και αλλιευτικά. Και η γαστρονομία μας είναι τμήμα του πολιτισμού που θέλουν να γνωρίσουν από πρώτο χέρι οι επισκέπτες και να το ζήσουν. Είναι ένας πολιτισμός πραγματικά στον οποίο πρέπει να ποντάρουμε. Έχουμε αυτές λοιπόν τις πολιτιστικές διαδρομές, το προσκύνημα του Αγίου Ιακώβου της Κοποστέλα, αλλά και άλλα που έχει χαρακτηρίσει την πολιτιστική κληρονομιά UNESCO. Έχουμε και ευρωπαϊκές πολιτισμικές διαδρομές που αναζητούν τον εμπλουτισμό, ε, τη διάδραση και την ε, ανταλλαγή. Και διευκολύνουν να σφυρατηθεί μια κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα. Από τις 24 διαδρομές ε, στην Ευρώπη έχουμε έξι. Ας πούμε τη μεγάλη διαδρομή πολιτιστική των Βίκινγκ, ε, την προϊστορική τέχνη, ε, οι αματικές πηγές, οι αματικές πόλεις και μια σειρά άλλες δράσεις. Η Ευρώπη θέλουμε να παραμείνει πρώτος προορισμός παγκοσμίω, γι' αυτό θα πρέπει να συνεργαστούμε και να δούμε τα στοιχεία που μας ενώνουν και τις πλατφόρμες που φέρνουν την Ευρώπη αντιμέτωπη με άλλες ε, περιφέρειες του κόσμου. Το 2018 θα είναι το έτος του τουρισμού Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας, μεγάλη ευκαιρία για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε και να γνωρίσουμε την κινέζικη αγορά. Μιλά, ας μιλήσουμε για το προσκύνημα του Αγίου Ιακώβου, ας μιλήσουμε για το δρόμο του μεταξιού, γιατί έτσι θα συνδεθεί η Ευρώπη με την Κίνα. Και θα πρέπει οι ροές να μην πηγαίνουν μόνο σε εμβληματικούς τόπους, αλλά και σε άλλους που είναι ενδιαφέροντες και έχουν λιγότερη συμφόρηση. Έτσι θα προχωρήσουμε με αηφορία, με ευθύνη αυτά μας εμπνέουν και θέλουμε ένα τουρισμό βιώσιμο, ανταγωνιστικό. Υπάρχει ένα μεγάλο δίκτυο. Είμαστε υπέρ των πλατφορμών ε, προβολής, γαστρονομία, πολιτισμός, ε, περιβάλλον, πολιτισμός σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Στη Γαλλικία ε, είναι πολιτιστικός ο τουρισμός και οι τουρίστες αυτοί αφήνουν 30% περισσότερο συνάλλαγμα και ως ε, προορισμός η Γαλλικία. Έχει γεματικές πηγές, έχει το δρόμο ε, ε, της Καμέλιας και έχουμε λουλούδια, φύση που μπορεί κάποιος να ανακαλύψει. Και αυτό δεν είναι εποχιακός τουρισμός. Έχουμε το Σαντιάγο de Κομποστέλα που διαχρονικά είναι φάρος στην Ευρώπη, αλλά θα πρέπει να αναπτύξουμε και τα άλλα πολιτιστικά μονοπάτια. Ευχαριστώ. Ja, Σας ευχαριστώ θερμά ε, για αυτές τις ε, ε πολυσχηδείς ε, ε παρουσιάσεις ε, τις οποίες ακούσαμε τα τελευταία μία, μία μισή ώρα. Έχουμε ξεπεράσει λίγο τον προβλεπόμενο χρόνο μας, αλλά νομίζω πως έχουμε άλλα 10 με 15 λεπτά για να μπορέσουμε να κάνουμε μία συζήτηση και θα ήθελα να ε, δώσω καταρχήν ε, το λόγο ε, στους συναδέλφους και συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια, οι οποίοι βρίσκονται σήμερα εδώ μαζί μας και τους οποίους καλωσορίζω θερμά. Οπότε σηκώστε το χέρι σας αν θέλετε να πάρετε το λόγο και ε, παρότι έχετε τις πινακίδες των ονομάτων σας ε, σας, όταν θα παίρνετε το λόγο ε, να μου λέτε ποιο είναι το όνομά σα, γιατί δεν μπορώ να τι διαβάσω, είναι μακριά αυτέ τι πινακίδε. Και σα παρακαλώ ο κάθε ένα να κάνει την παρέμβασή του για όχι παραπάνω από ένα λεπτό. Εδώ η κυρία ε, μπροστά μου την είδα πρώτη, οπότε. Καφαντάρη Χαρά από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, από την Ελλάδα. Ε, ο τουρισμός αποτελεί δραστηριότητα μεγάλης σπουδαιότητα της ελληνικής και της ευρωπαϊκής οικονομίας και μοχλό ανάπτυξης. Στην Ελλάδα ο τουρισμός συνεισφέρει ε, σημαντικά στην οικονομία και αποτελεί βασικό πυλώνα της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Στη χώρα μας, στις 16 Μαΐου του 2016, πραγματοποιήθηκε στο Κοινοβούλιο δεύτερη Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Διάσκεψη για τον Τουρισμό με συμμετοχές 16 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ένωση Μεσογειακών Λιμένων Κρουαζιέρας, Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού και ΟΟΣΑ. Ο τουρισμός λοιπόν είναι τρόπος προσέγγισης των λαών, των πολιτισμών, των αντιλήψεων και φέρνει σημαντικά οικονομικά ωφέλη. Η Ελλάδα προσφέρει πλούσιο τουριστικό προϊόν, προωθεί δυναμικά το θεματικό τουρισμό σαν στρατηγικό άξονα της εθνικής τουριστικής πολιτικής. Προωθούμε τον πολιτιστικό τουρισμό, θρησκευτικό, υγείας, ιαματικό, αθλητικό, τουρισμό πόλεως αλλά το ζητούμενο δεν είναι μόνο η ανάπτυξη του εσωτερικού τουρισμού όπως ελέγχθη εδώ εντός της Ευρώπης και μόνο, αλλά και η προώθηση της Ευρώπης σαν πρώτο τουριστικό προορισμό για τρίτες χώρες. Εδώ θα αναφέρω ότι πρόσφατα υπογράφτηκε στις 19 Σεπτεμβρίου στη Μόσχα η έναρξη του έτους τουρισμού Ελλάδας-Ρωσίας που θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του 2018 ενώ όπως ελέγχθη το έτος 2018 είχε ανακηρυχθεί έτος τουρισμού Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας. Ε, η Ευρώπη με την ιστορική και πολιτιστική της παράδοση παραμένει ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο, ωστόσο μπορεί να αυξήσει κατά πολύ ακόμα την επισκεψιμότητά της και από τρίτες χώρες. Η συνεργασία των κρατών, των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των λαών είναι καθοριστική ώστε πραγματικά η Ευρώπη να είναι ο πρώτος τουριστικός προορισμός. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπω ένα πρόσωπο του Βελτικού. Πιέτρο Σάλα, από την Ιταλία θέλω να σας γνωστοποιήσω αυτό το δίκτυο που είναι μουσεία και επιχειρήσεις πάνω από 60 μουσεία συμμετέχουν και μεγάλες, ε, πιο μεγάλες ιταλικές επιχειρήσεις από τη μόδα, από η Φεραγκάμου, το design όπως λέει και διάφορες μάρκες τροφίμων όπως η Μπαρίλα, η Περόνη συμμετέχουν, η Καμπάρη, η Μαρτίνη. Είναι ένα δίκτυο που ε, ε, καλύπτει όλη την επικράτεια και προσφέρει αυτή την πολυσχηδή προσέγγιση, το βιομηχανικό τουρισμό που πάνω απ' όλα για έναν κόσμο ε, ε, ε, τουριστών που καταφθάνουν πολύ μακριά, όπως είναι οι Κινέζοι τουρίστες. Οι Κινέζοι τουρίστες πραγματικά έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά ζωντανά τις μεγάλες επιχειρήσεις, τις μεγάλες μάρκες ιταλικές και είναι μουσεία που δεν χρειάζονται εξηγήσει. Είναι μουσεία που άμεσα εμφανίζονται, προέρχονται από τους ανθρώπους από τα μουσεία. Βιομηχανία, μουσεία. Ας πούμε, έχουμε μια μάδα μουσείων στη Ρωμάνια που είναι η μεσαία της γης των κινητήρων που εκεί είναι μουσεία που αφορούν τις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες Ιταλίας με εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο και πιστεύουμε ότι πραγματικά μπορούν να αποτελέσουν ένα δίκτυο, έναν προορισμό κάπως διαφορετικό που όμως αντιπροσωπεύει στον αλλοδαπό, στον τουρίστα που έρχεται από μακριά μια εικόνα για την Ιταλία θετική, παραγωγική με μάρκες που είναι πάρα πολύ γνωστές, πασίγνωστες. Σας ευχαριστώ θερμά. Δεν βλέπω να ζητάει κάποιος άλλο το λόγο. Άλλωστε ήταν και πολύ μακρά η συνεδρία σήμερα, πολλές ομιλίες η μία μετά την άλλη, πολλές συζητήσεις, οπότε νομίζω πως θα μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε κάπου εδώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμότατα όλους τους συμμετέχοντες σήμερα εδώ και τις παρεμβάσεις τους. Νομίζω πως ε, όλες αυτές τις προσκλήσεις που ακούσαμε για τις διάφορες περιοχές της Ευρώπης αλλά και για την Κίνα ε, δεν θα προλάβουμε να ανταποκριθούμε σε όλες αυτές ε, γιατί αυτό θα σημαίνει ότι θα πρέπει να ταξιδεύουμε όλη την ώρα κάτι που θα μας ευχαριστούσε βέβαια πολύ αλλά δεν είναι δυνατόν. Πάντως σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σίγουρα τη μία ή την άλλη περιοχή κάποια στιγμή θα την επισκεφτούμε, θα ταξιδέψουμε εκεί. Ε, ελπίζω όλοι σας να είχατε τη δυνατότητα να σχηματίσετε μια εντύπωση της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς που έχει να προσφέρει η Ευρώπη, ειδικότερα όσοι έχετε έρθει από μακριά, και ίσως και οι Βρυξέλλες, ίσως δηλαδή να είχατε δυνατότητα να απολαύσετε λίγο τις Βρυξέλλες εδώ στην επίσκεψή σας. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους θερμότατα για τη συμμετοχή σας σε αυτή τη διάσκεψη και απλώς να σας ενημερώσω και να σας ε, καλωσορίσω σε μια μικρή δεξίωση η οποία θα λάβει η χώρα στο εστιατόριο των μελών του Κοινοβουλίου, δηλαδή μόλις βγείτε εδώ από την αίθουσα, θα περάσετε την Πασαρέλα και θα κατεβείτε στο άλλο λοιπόν κτίριο, το δίπλα κτίριο, στο Εσόγειο. Εκεί ελπίζω ότι θα μπορέσετε λοιπόν να βρείτε το που λαμβάνει η χώρα. Ε, αν δεν το βρείτε, ρωτήστε κάποιον, ίσως να υπάρχουν και κάποιες πινακίδες εκεί. Σας ευχαριστώ και πάλι όλους εδώ για τις παρεμβάσεις σας και σας εύχομαι καλό βράδυ σε όλους. Ευχαριστώ πολύ.